liebe kolleginnen und kollegen! ich störe ungern die fröhliche vorweihnachtslaune. Ε, τώρα δεν θέλω και εγώ να σας βγάζω από τη ραστόνη, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να καλωσορίσουμε και τα μέλη της Επιτροπής Προπολογισμού. Είναι μεγάλη μας τιμή να δεχόμαστε εδώ πέρα τόσο εξέχοντες συναδέλφους όπως τον κύριο Μπέγκε, την κυρία Χάουγ γιατί έχουμε να συζητήσουμε ένα δύσκολο θέμα στην κοινή συνεδρίαση. Είναι ο πρότυπος μεσονομικός κανονισμός για ΣΔΙΤ, για πράξεις κατεξιοδότηση. Τώρα θα μιλήσω αγγλικά, γιατί το έγγραφο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι στα αγγλικά. Οπότε, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 η Κομισιόν υιοθέτησε έναν κανονι... πρότυπο κανονισμό για ΣΔΙΤ σύμφωνα με το άρθρο 209 του κανονισμού που προβλέπει πως οι συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα θα λαμβάνουν μια έμεση απαλλαγή από την ε, Κομισιόν. Έτσι αλλάζει η πάγια πρακτική που γίνεται σε κάθε κοινή επιχείρηση και ΣΔΙΤ για να γίνεται η απαλλαγή ε, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση για να διατηρηθεί η διαφάνεια. Συμβούλιο και Κοινοβούλιο βεβαίως μπορούν να έχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις στην όλη διαδικασία, καθώς ο νέος κανονισμός ο οποίος ιδιοθετήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού. Οποιαδήποτε απόφαση αφορά την ε, εξέταση των πράξεων αυτών κατεξιοδότης θα πρέπει να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία. Οι συνεισηγητές, η κυρία Κρέσλε και ο κύριος Ριβελίνη προτείνουν στις επιτροπές μας να γύρουν ένσταση στον κανονισμό για τον ε, πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τη ΣΔΙΤ και να προτείνει στην Κομισιό να επανεξετάσει την απαλλαγή. Στην κοινή μας συνεδρίαση της 6 Νοεμβρίου αποφασίσαμε να ζητήσουμε η περίοδος εξέτασης να παραταθεί και το Κοινοβούλιο πρέπει να λάβει μια απόφαση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2014. Το σχέδιο ψηφίσματος για την ένσταση αυτή στα λίστα μέλη των Επιτροπών μέχρι στις 4 Δεκεμβρίου μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου δεν είχαμε τροπολογίες και εν τω μεταξύ έχουν προταθεί τα εξή. Πρώτα απ' όλα, μια ενδιάμεση λύση να υπάρξουν παρεκκλήσεις για κάθε μία από τις ε, βασικές πράξεις και τους ε, ανάλογους ε, εσωτερικούς ε, κανονισμούς. Προετοιμάζουν οι συνάδελφοι της ήτρε τις ανάλογες τροπολογίες. Αργότερα το 2014 η Κομισιόν θα προτείνει μία μόνιμη λύση, μία τροποποίηση του ίδιου του κανονισμού και κατόπιν έναν κανονισμό κάτω εξουσιοδότηση έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί και το πλαίσιο των ΣΔΙΤ με αυτά τα οποία θα ισχύσουν με τον ε, κανονισμό GDI. Εμείς θεωρούμε και η συγκίτρια θεωρεί πως ε, έχουμε εδώ πέρα ένα καλό συμβασμό και τώρα βεβαίως μπορεί να πρέπει να συμφωνήσει Συμβούλιο Κοινοβούλιο και Κομισιόν με κάποιες ε, κοινέ δηλώσεις. Χθε είχαμε κάποια πάρα πολύ θετικά μηνύματα από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει πέρσι 8 Ιανουαρίου. Παρ' όλα αυτά, αυτή την ώρα, οι συνεισηγητές προτείνουν να συνεχίσουμε την διαδικασία της ένστασης στον κανονισμό κατεξιοδότηση και άρα να υπερψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος, δηλαδή ε, την ένσταση. Οι συνεισηγητέ βεβαίω είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν την διαδικασία μέσω μια τροπολογίας στην Ολομέλεια μόλις το Συμβούλιο εγκρίνει τι κοινέ δηλώσει. Ωραία. Νομίζω περιέγραψα την κατάσταση, την διαδικασία δηλαδή, οπότε θα ήθελα τώρα να ρωτήσω εάν οι δύο συνεισηγητέ ε, θέλουν το λόγο των συνεισηγητή, δηλαδή τον ιδέα, κυρία Γκρέσλε. Χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Πρέπει να βοηθήσουμε λίγο την Κορεπέρ να λάβει την απόφασή της στις 8 Ιανουαρίου. Εάν είναι διατεθειμένο το Συμβούλιο να αναλάβει την ε, άμεση απαλλαγή σε μια απόφαση, τότε θα φροντίσουμε να ανακαλέσουμε την σημερινή μας απόφαση στην Ολομέλεια. Οπότε, μία μεταβατική λύση έχουμε εδώ πέρα. Όπως είπα. Και αν τα δεχτεί αυτά το Συμβούλιο στις 8 ε, Ιανουαρίου, το σε όλες Κομισιόν θα προτείνει μία λύση κατά αποκοπήν σύμφωνα με το άρθρο 209. Είναι μία διαδικασία όπως είπα για να ασχίσουμε λίγη πίεση είναι ένα προληπτικό μέτρο αν θέλετε το οποίο μπορεί να ανακληθεί Βεβαίω ξέρουμε τους φίλους μας στο Συμβούλιο καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί ελπίζω αυτή η ανακοχή χριστουγεννιάτικη να διατηρηθεί αυτά αλλιώς τι να πω, αν δεν τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ, εμπασφέρτως. Ναι, ε, ίσως να είναι τόσο πολύπλοκος αυτός ο κανονισμός να μας κάνει να, να σκεφτούμε το να αλλάξουμε δουλειά. Αστείευομαι βεβαίως, λέει ο πρόεδρος. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση, αλλά βεβαίως υπάρχει μια παράληψη που πρέπει να διορθωθεί υπάρχουν οι δύο πραγματευτές αλλά και ε, βεβαίως ε, άλλα εξέχοντα μέλη εδώ πέρα. Οπότε ζητώ συγγνώμη που δεν χαιρέτησα προσωπικά διασημότητες όπως την κυρία Τρότμαν. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, παρουσία σας. Λοιπόν, ο κύριος Μίλντερ έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ δυσκολεύομαι και είναι λιγάκι περίεργο όταν η Επιτροπή κάνει ακριβώ αυτό που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, εμεί να υπαναχωρούμε. Αλλά το γεγονό ότι είναι και μα ε, διαβεβαιώνει ότι ε, θα ακολουθηθεί η συμφωνία με το Συμβουλίο, ακολουθώντα και το πνεύμα των Χριστουγέννων, θα συμφωνήσω με την πρόταση τη συγκητρία. Ωραία, υπάρχουν άλλοι συναδέλφοι που θα ήθελαν το λόγο. Κύριε Οντή. Ευχαριστώ. Σίγουρα δεν θα εκπλαγείτε που και εγώ θα υποστηρίξω τη στρατηγική της ΙΝΚΕ, έχει δίκιο. Γιατί αυτό το ζήτημα το Συμβούλιο θα κάνει ό,τι θέλει, αλλά από την πλευρά μου θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή γιατί η Επιτροπή θα μπορούσε, θα μπορούσε να έχει συνεχίσει με τη δικιά της πρόταση, στην οποία περίπτωση θα έχει λιγότερη σημασία ψήφος, αλλά ε, ε, το σημαντικό είναι που θα παραμείνει η απαλλαγή στα χέρια του Κοινοβουλίου. Η απαλλαγή δεν είναι απλώς μια αποδοχή των λογιστικών καταστάσεων. Υπάρχει επίσης και ένας πολιτικός έλεγχος Υπάρχει επίση ένα στοιχείο καινούριο στη, διαδικασία αυτή που είναι οι ηλεκτρονικέ παραγγελίε και εδώ πειραματιζόμαστε. Επομένω είναι σημαντικό ο πολιτικό ρόλο που αναλαμβάνει το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία λήψη απόφαση, σε αυτή την αλυσίδα. Ειδικά για τον συγκεκριμένο κανονισμό που αναφέρεται στι ΔΙΤ. Το άρθρο 29 δεν διαθέτει το κείμενο, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, Διαφορετική διαδικασία. Η πολυπλοκότητα και η γραφειοκρατία δεν προέρχεται από τη διαδικασία της απαλλαγής. Αυτή τη στιγμή στο λεκτικό συμβούλιο κάνει την, συνέδριο κάνει τη δουλειά του, η διαδικασία της απαλλαγής είναι πάρα πολύ γρήγορη. Στην πραγματικότητα η γραφειοκρατία προέρχεται από τους κανονισμούς που αφορούν στη δημόσια λογιστική. συζητώντας με διευθυντές, με διευθυντικά στελέχη ε, που συμμετέχουν στις ΔΙΤ, ζητούν απλοποίηση. Και βεβαίως θέλουν να τηρήσουν τους κανόνες ε, της, ε, των δημοσίων προεπιμήθειών και τα λοιπά και τους κανόνες της διαφάνειας, αλλά αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλοποιημένοι. Και αναρωτιέμαι λοιπόν αν συμφωνεί και συνάδελφοι, ότι ο νέος ε, δημοσιονομικός κανονισμός χωρίς την πραγματικότητα να υπονομεύει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, παρόλα αυτά ακολουθεί διαδικασίε οι οποίε ταιριάζουν με τι γενικότερε διαδικασίε των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επομένω, αναρωτιέμαι αν πραγματικά έχουμε καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω μια επιθυμία. Όπως ξέρετε, αυτές οι τελικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου τομέα και ιδιωτικού είναι πάρα πολύ σημαντικά στα πλαίσια του 2020, του Horizon 2020, ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που εμπεριέχει τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις, συμμετοχή επιχειρήσεων και βεβαίως Χρειαζόμαστε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα για να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Και με έναν απλό τρόπο, με έναν ομαλό τρόπο στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και θεωρώ ότι αυτό που ψηφίζουμε σήμερα μας οδηγεί ακριβώς στο να επιτύχουμε κάτι τέτοιο και Ήδη από το 2014 ξεκινάει αυτή η πορεία προς το 2020 χωρίς να δημιουργούμε επιπλέον εμπόδια για τους επιχειρηματίες της Ευρώπης και τους ε, ερευνητές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η Επιτροπή. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως συμφωνούμε με τους εισηγητές. Κάποιοι δεν εκφράστηκαν ακόμα, δεν έχει γνωμοποιήσει η Επιτροπή Ήτρε. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι όλοι συμφωνούν πως θα πρέπει να επιτύχουμε μια απλοποίηση των κανόνων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις καθώς και τις διαδικασίες απαλλαγής. Και Εξού και θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία με το Συμβούλιο. Συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα για να τους οδηγήσουμε προς τη στήριξη αυτής της κοινή δήλωσης. Ελπίζω μετά τη συνάντηση της 8ης Ιανουαρίου στο Κορεπέρ και αυτής που θα έλεγε χώρα σε 9 Ιανουαρίου θα μπορέσουμε να στήριξουμε όλοι από κοινού αυτήν την ε, κοινή δήλωση και ελπίζω επίσης να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Κύριο Ντί, θα απαντήσω σε αυτά που είπατε λέγοντας ότι όσον αφορά την κάτι της υπάρξης που βασίζεται στο άρθρο 209, ο σκοπός μας είναι η απλοποίηση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Πρώτον, δημοσιονομικός σχεδιασμός, απλοποιημένος απλοποιημένη διαδικασία για την έγκριση του προϋπολογισμού καθώς και για τον πίνακα του προσωπικού καθώς και για τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία κάποιων συναλλαγών αλλά και βεβαίως τα λογιστικά πρότυπα που θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα διεθνή ε, λογιστικά πρότυπα. Απλοποίηση λοιπόν για αυτήν την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά σε καμία περίπτωση μην, μπορεί, μην φανταστείτε ότι θα υπάρξει ξεχωριστή απαλλαγή. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να γίνει στην ε, αναθεώρηση που όπως είπε η συγγήτρια θα λάβει χώρα σε ένα χρόνο. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να ζητάει το λόγο. Λέει ο Πρόεδρος μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε με ηλεκτρονικό τρόπο θα ψηφίσουμε. Ναι. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Πόσοι είναι παρόντες, πόσοι ψηφίζουν. Αρχή της ψηφοφορίας. Βλέπω εδώ ότι οι φιλελεύθεροι είναι υπεράριθμοι. Άρα μπορώ εγώ να μην ψηφίσω, να απέχω. Να μην ψηφίσω ούτε εγώ ούτε άλλοι δύο. Ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία. Ακυρώστε το αποτέλεσμα. Αρχή της ψηφοφορίας εκ νέου. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Ωραία. Οι δύο λοιπόν επιτροπές ψήφισαν ομόφωνα υποστηρίζοντας την πρόταση των εισηγητών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απολύτως σαφές το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και σας εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλή αντάμωση τον καινούριο χρόνο. Παρακαλώ, όσοι είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, μπορείτε να παραμείνετε στην αίθουσα και θα συνεχίσουμε. Ολοκληρώθηκε η κοινή μας συνεδρίαση, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και κατόπιν θα συνεχίσει η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού.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 μπορούσα να διαλέξω Μόλις με ενημέρωσαν πως ο κύριος Μαρινέσκου βρίσκεται στην Επιτροπή Μεταφορών σε κάποια ψηφοφορία, οπότε προτείνω να επαναλάβουμε την συνεδρίαση για να περάσουμε σημείο 14 την έκθεση Bart τη της ημερήσιας διάταξης. Νομίζω αφορά την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Καλωσορίζω τον κύριο Βέσμπεργκ του Ενεκτικού Συνεδρίου. εκπροσώπους της Κομισιόν βεβαίως δεν έχει νόημα η συζήτηση, οπότε θα περιμένουμε να σχέδιο.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 So, um, one question to our colleagues from EPP. Do you Να ρωτήσω τους συναδέλφους του ΕΛΚ. Ε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και να έρθει μετά ο εισηγητής. Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση με λίγα λεπτά καθυστέρηση καλωσορίζω από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τον κύριο Βέρνερ Χόιερ, τον Γενικό Διευθυντή. Καλώς ήρθατε. Προτείνω να ξεκινήσουμε αμέσως. Θέλει κάποιο από το ελεγκτικό συνέδριο τον λόγο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όχι. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με εσά και μετά θα περάσουμε στην ετήσια έκθεση, στα κομμάτια δηλαδή τα οποία οφείλει να δώσει απαλλαγή το Κοινοβουλίο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που δίνεται στην τράπεζά μας, τραπεζά σας αν θέλετε, την δυνατότητα να σας εξηγήσουμε, να σας δώσουμε κάποιες πληροφορίες περισσότερες στην συνάντηση της Επιτροπής σας. Πρώτα απ' όλα, όπως ήδη ανέφερθηκε και από τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, πριν από ένα μήνα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θεωρεί ότι είναι αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Και εστιάζουμε ιδιαίτερα, όπως μας έχει ζητηθεί, στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Όπως θα γνωρίζετε, ενημερώσαμε το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο τον Οκτώβριο για τις πρωτοβουλίες που είχαμε αναλάβει έως τότε και τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Δύο θέματα τονίστηκαν και από πολλούς από εσάς τους ευρωβουλευτές ήταν το ζήτημα της απασχόλησης, το ζήτημα των δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της τραγικής κατάστασης όσον αφορά την ενεργεία των νέων σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δημιουργήσαμε ένα ποσό ε, δεσμευμένο για 6 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την καταπολέμηση ε, των, ε, ε, αυτής της ανεργίας των νέων μέσω δανείων. Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες που έχουν τη μερίδα του λέοντος στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Ο στόχος μας είναι η ανεδότηση με 18 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και σε αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί το EIF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Επενδύσεων. Συνολικά φτάνουμε στα 21 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα επενδυθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη χρονιά, αυτό το έτος. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την συμμετοχή της τράπεζας μας στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν μέρος των διαρθρωτικών ταμείων ε, του χρόνου και τα επόμενα χρόνια, αν χρειαστεί, αρχικά ως εργαλείο ε, εγκυοδοσίας για να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε από τα κράτη-μέλη να μας δώσουν το πράσινο φως και να μας πούν ε, σε ποιο βαθμό επιθυμούν να συμμετάσχουν. Πάντως το πρόγραμμα αυτό έχει συζητηθεί διεξογικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και συζητήσαμε διάφορες επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας για τη βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης υπάρχει το ζήτημα το χρηματοδότηση της στρατηγικής για 2020 και το ζήτημα των ιδίων πόρων. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας όλο το έργο που αφορά στην εξωτερική διάσταση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου το 10% της δανειοδότησης ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων απευθύνεται προς ε, χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκουμε η δανειοδότηση αυτή να ευθυγραμμίζεται με τους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμπεριλαμβάνουν την ενίσχυση της σταθερότητας, την ενίσχυση της ποιότητας της διακυβέρνησης σε ορισμένες χώρες ή επίσης ε, σε επενδύσεις για την καταπολέμηση της ε, αλλαγής του κλίματος. Και κοιτώντα σας κύριε Κάλφιν το, το, το ε, θυμούμε ακόμα περισσότερο γιατί είμαστε ευγνώμονες για την μεγάλη υποστήριξη που είχαμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο των επενδύσεων ε, υψηλό όπως και στο παρελθόν και νομίζω ότι βρισκόμαστε, κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε για τη βοήθεια που μας δώσατε. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο για να μην μακρηγορήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah, thank you very much, uh, Mr. Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Κνάπεν. Ήσασταν συνοπτικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχουν οι βουλευτές. Ο εισηγητής μας βεβαίως δεν έχει έρθει ακόμα. Οπότε θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Κύριε Κάλβιν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποια σχόλια στην έκθεση Μαρινέσκου πριν έρθει και μετά εγώ θα φύγω δυστυχώς, δεν θα συναντηθούμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Κνάπε. Αν δεν το ξέρετε οριστικοποιήθηκαν οι τριμερείς διάλογοι και τώρα έχουμε μια τεχνική διαδικασία για να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός, κάτι το είναι θετικό και για εμάς και για όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται η τράπεζα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που περιέχονται στην έκθεση που ενδιαφέρουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσω με αυτό το οποίο είπε ο κ. Κνάπεν για τη δουλειά που κάνει η τράπεζα με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάτι σχετικά νέο για την τράπεζα. Τη συζήτησε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο να αφιερώσει κάποια κονδύλια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω πως ε, ήδη έχουμε κάποια αποτελέσματα στις ε, παραγράφους 45 έως 47 της έκθεσης ε, ο κύριος Μαρινέσκου προτείνει να περάσουμε στα κριτήρια επιλεξιμότητας και να δούμε με βάση ποιες αρχές η χρηματοδότηση των τραπεζών φτάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται κυρίως μέσω ενδιαμέσων βεβαίω. Τώρα χωρίς να πάμε στα συγκεκριμένα κριτήρια επιλεξιμότητας, ίσως όταν αποκτηθεί κάποια εμπειρία η τράπεζα μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των δανείων, εάν είναι πιο αποτελεσματικά, εάν μεταφέρουν αυτή την ευκολία της εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση στους τελικούς δικαιούχους κτλ. Κάποια αξιολόγηση δηλαδή για το εάν αξίζει να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία και αν υπάρχουν κάποιες ε, ιδέες για αλλαγές. Στην παράγραφο 60 ο εισηγητής λέει πως πρέπει να γίνει μια ειδική έκθεση, να ζητήσουμε δηλαδή μια έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο για τις, ε, τον εξωτερικό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κοιτάξτε, Υπάρχουν πολλές σχετικές πληροφορίες και έρευνες, αλλά οπωσδήποτε μία έκθεση από το ελεγκτικό συνέδριο είναι καλή ιδέα. Ίσως θα έπρεπε να συμπέσει με την ενδιάμεση αναθεώρηση που προβλέπεται για το 2016-2017, έτσι ώστε να δούμε τα ευρήματα όταν θα συζητήσουμε ξανά την εντολή. Μετά, στην έκθεση ζητείτε να αυξηθούν τα μέσα με τα οποία μοιράζεται ο κίνδυνος. Πρέπει να φροντίσουμε βεβαίως να μην εμπλακούμε σε καθαρά τραπεζικές αποφάσεις της τράπεζας. Και ένα βασικό κριτήριο θα πρέπει να είναι η διακριτική ευχέρεια της τράπεζας για να μπορεί να λειτουργεί και να έχει πρόσβαση σε φθηνά κονδύλια. Εγώ δεν θα ήθελα το Κοινοβούλιο να κρίνει την αύξηση ή τη μείωση του κινδύνου που αναλαμβάνει η τράπεζα. Κάτι άλλο που είναι επίσης ενδιαφέρον για τη δουλειά μας και αφορά το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προπολογισμό της Ένωσης είναι όλα αυτά τα μέσα που στόχο έχουν να συμπληρώσουν την, ε, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην Επιτροπή Προπολογισμού πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Είχαμε και κάποιες ακροάσεις, μελέτες κτλ. Ε, κτλ αλλά κοιτώντας τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές νομίζω πως από καιρού καιρόν καλή ιδέα θα είναι να δούμε πώς θα μπορούσε η τράπεζα να βοηθήσει τους δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν καλύτερα την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία όπως ξέρουμε θα είναι επενιχρή. Εγώ δεν θεωρώ πως η τράπεζα μπορεί να αντικαταστήσει τα ευρωπαϊκά ταμεία, γιατί είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεν δίνει επιχορηγήσεις, αλλά σε συνδυασμό με τις επιχορηγήσεις νομίζω μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Τέλος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα μια επιτροπή σοφών υπό την προεδρία του Μισελ Καμπτεσίου με στόχο να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα για να συναντηθούν. Ξεκινήσει να λειτουργεί και Νομίζω πως έχουμε κάποια θετικά μηνύματα. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να αξιολογήσουμε τη λειτουργία. Υπάρχει επίσης τεράστια διαφωνία από την πλευρά των ΜΚΟ. Λένε πως δεν είναι πλέον ε, διαφανής η λειτουργία, αλλά είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια ισορροπία και να δούμε αν πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, την κοινή χρηματοδότηση με άλλα ιδρύματα και αν πρέπει να υπάρχει αυτή η πλατφόρμα που ξεκίνησε προσφάτως. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Επιτροπή Εσωτερική Αγοράς προσπαθούμε να στηρίξουμε την πολιτική χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και το πρώτο που ήθελα να πω, το ανέφερε και ο κύριος Κάλφιν. Πώς σκοπεύετε να οργανωθείτε, θα δίνετε η χρηματοδότηση κατευθείαν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή προτίθεστε να περάσετε από τα δίκτυα, τα τραπεζικά σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε γιατί θέλουμε να το ανακοινώσουμε και στις ε, χώρες μας. Στην ε, Γερμανία αλλά και σε πολλές χώρες έχουμε θέμα ρευτότητας όπως ξέρετε. Πρώτη ερώτηση λοιπόν. Πώς ε, πρόκειται να οργανωθείτε. Ξέρω ότι κάτι θα έχετε ήδη προβλέψει και εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Επίσης δεύτερον, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της καινοτομίας και της έρευνας. Βοηθάτε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα παραδείγματο χάρη συνεργασία με Ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα σε τοπικό επίπεδο. Γιατί βεβαίω οι μεγάλε επιχειρήσει, οι όμιλοι επιχειρήσεων, οι πολυεθνικέ έχουν δικά του τμήματα ερευνητικά. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πολλές φορές πολύ περισσότερο στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας. Αν μπορούμε λοιπόν να τους βοηθήσουμε, θα ήταν εξαιρετική ιδέα. Μπορείτε να μας πείτε. Γιατί εμένα θα με ενδιέφερε στην εκλογική μου περιφέρεια να το ανακοινώσω αν υπάρχει κάτι. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ καλό, όχι μόνο για τα Χριστούγεννα, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο νέο. Κύριε Κνάπεν, θέλετε να απαντήσετε τώρα. Έχω και τον κύριο Οντί, ο οποίος θέλει να κάνει ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα στοιχεία που μας δώσατε. Ήταν πολύ ενημερωτικά. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το κοινωνικό κεφάλαιο. Είδαμε ότι κάποιες κυβερνήσεις προτείνουν αύξηση κεφαλαίου της άξιος των 10 δις, που σημαίνει χρηματοδότηση που θα φτάσει μέχρι τα 60 δις. Αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των 10 δις που προκαλεί, ε, μάλλον οδηγεί σε μία χρηματοδότηση επιπλέον της τάξης των 60 και τα 120 δις που ήδη έχουν ε, δεσμευθεί τα κράτη-μέλη να δώσουν. Γιατί δεν αφήνουν, αν θέλετε, ε, αυτά τα υπόλοιπα χρήματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή 220, 220 δισεκατομμύρια τα οποία ουσιαστικά παραμένουν ε, δεσμευμένα γιατί από τη μία έχουμε τα 10 δις τα οποία οδηγούν σε μια χρηματοδότηση 6 εξαπλάσια, 60 δις και από την άλλη ε, δεν βλέπω το συσχετισμό μεταξύ των 220 δισεκατομμυρίων που ακόμα πρέπει να ελευθερωθούν από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, εδώ και έξι χρόνια περίπου το Κοινοβούλιο ζητάει την εποπτεία της τράπεζάς σας. Και αυτό δεν γίνεται. Στην αρχή μας είχαν πει ότι όλες οι τράπεζες επενδύσεων, μακροχρόνων επενδύσεων, δεν είναι αντικείμενα εποπτείας. Μάλιστα Είχαμε ζητήσει από τον Υπουργό τον πρώην Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας που σήμερα είναι επικεφαλής του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, ο οποίος απάντησε ότι αυτό δεν ήταν ε, κάτι που κανονικά έπρεπε να απαγορεύεται. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραμένει χωρίς ε, απολύτως καμία εποπτεία. Η Τραπεζική Ένωση η αρχή εποπτεία του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη, έχει κάνει διάφορες προτάσεις και τελικά βλέπουμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζάς δεν ακούει. Δεν ανταποκρίνεται. Δεν ξέρω αν οι διοικητές που είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουν να κάνουν κάτι. Μη μου απαντήσετε εδώ ότι υπάρχει συμφωνία με την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου. Επί έξι χρόνια την ακούω αυτή την απάντηση. Επίσης, η τράπεζά σας προτίθεται να υποβάλει τα σημεία που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του προγράμματός της στους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών μας. Άλλη ερώτηση όσον αφορά τις ε, μακροχρόνιες ε, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ είχα βρει την ιδέα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα να συνεργαστείτε με ειδικού του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ξέρω βεβαίως ότι έχετε πολλούς εμπειρογνώμονες, αλλά πώς βλέπετε μια πιθανή συνεργασία για τους τομείς παραδείγματος χάνει της ενέργειας, των μεταφορών, για μια τέτοια συνεργασία. Ξεκινήσατε σήμερα τις δηλώσεις σας λέγοντας θα μιλήσω για την τράπεζά σας. Ναι, όντως πρόκειται για την τράπεζα των κυβερνήσεων. Το Κοινοβούλιο έχει προτείνει εδώ και πολλά χρόνια να υπάρξει κάποιος τρόπος συνεργασίας σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τράπεζας. Το είχαμε προτείνει. Πώς σας φαίνεται η ιδέα αυτή να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδεδεμένο μέλος ή μέλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήσεις που μου κάνετε, για τις παρατηρήσεις σας. Ας ξεκινήσω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δύο-τρία σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο αναγνωρίστηκε στο σεμινάριο που διοργάνωσε η Fitch πριν λίγες ημέρες στο Λονδίνο έχει σχέση με την έλλειψη ζήτησης. το οποίο προφανώ έχει σχέση με την κατάσταση τη οικονομία. Εάν υπάρχει ανάπτυξη, αν υπάρχει στασιμότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στασιμότητα αλλά επίσης και κάτι που συνδέεται με την ε, παρατηρήση του κυρίου Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είμαστε, οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά εξαρτημένες από την δανειοδότηση από τις τράπεζες, εάν συγκριθούμε με τις ΗΠΑ. Δηλαδή οι επιχειρήσεις ε, βασίζονται στο κατά 80% στη χρηματοδότηση από τη, τον τραπεζικό τομέα. Και μόνο ε, και για το ποσοστό το οποίο προέρχεται από μετοχικό κεφάλαιο είναι πολύ μικρότερο. Αυτό είναι ακριβώ το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει στι ΗΠΑ, όπου εκεί οι επιχειρήσει είναι πολύ λιγότερο εξαρτώμενε από τι τράπεζε. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μα είναι ότι όταν μια επιχείρηση εξαρτάται τόσο πολύ από την, από την τράπεζα και όταν ταυτόχρονα ασκούνται σοβαρέ πιέσει στι τράπεζε που πρέπει να συρρυκνώσουν τι δραστηριότητέ του προκειμένου να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους, να μειώσουν το ρίσκο τους ή επίσης να ακολουθήσουν τους νέους κανονισμούς της νέα νομοθεσία όπως για παράδειγμα τη φεραγγιότητα 3 αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις επιχειρήσεις που χρειάζονται χρήματα. Και αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο που συμβάλλει στην κρίση την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη μαζί με τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Αν έχουμε μια επιχείρηση στην Ιταλία, μια μικρομεσαία επιχείρηση στην Ιταλία και στην Αυστρία, ο τρόπο με τον οποίο θα αναζητήσει τραπεζική χρηματοδότηση είναι τελείω διαφορετικό γιατί το spread υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επιτόκιο δανειοδότηση από τη μια χώρα στην άλλη. Και αυτή η κατάσταση υπονομεύει τι δραστηριότητε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν με ρωτάτε θα οργανωθούμε. Όπως γνωρίζετε εμείς δεν, είμαστε τράπεζα λιανικής, δεν έχουμε ATM. Επομένως θα χρησιμοποιήσουμε το τραπεζικό δίκτυο των τραπεζών ε, που έχουν τέτοιο ε, δίκτυο λιανικής στα κράτη-μέλη. Εκείνοι γνωρίζουν τους πελάτες τους, εκείνοι γνωρίζουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες, εκείνοι είναι σε καλύτερη θέση να κρίνουν. Και έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα κινηθεί μέσω αυτών των ε, τοπικών τραπεζών. Έχουμε ήδη ξεκινήσει ένα πρόγραμμα στην Ελλάδα, λίγο πριν το καλοκαίρι. Δύο προγράμματα μάλιστα. Πρώτα απ' όλα ένα σύστημα αγκαιοδοσία για τι ε, μικρομεσαίε επιχειρήσει, για την ακρίβεια για τι τράπεζε οι οποίε δανείζουν σε μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και δεύτερο, ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο δεν εντάσσεται ακριβώς στις ε, κύριε δραστηριότητε μα, αλλά ήταν απολύτως απαραίτητο που ήταν η χρηματοδότηση του εμπορίου, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο στην Ελλάδα. Μια εγγυητική επιστολή. Κάτι τόσο απλό, απολύτω απαραίτητο για την καθημερινή λειτουργία της οικονομίας. Ξεκινάμε ένα παρόμοιο πρόγραμμα στην Κύπρο. Ένα σύστημα εγκυοδοσίας πρώτα απ' όλα. Στην Πορτογαλία. και θα αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα καθώς αυτά ανακύπτουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Φυσικά αυτή η προσέγγιση ενέχει κινδύνους. Έναν απλό κίνδυνο θα σας αναφέρω. Αυτή τη στιγμή οι Υπουργοί Οικονομικών στο πλαίσιο της συζήτησης για την Τραπεζική Ένωση συζητούν το ενδεχόμενο του Μπέιλιν, in κουρέματος των καταθέσεων. Εάν εμείς έχουμε ένα όγκο πιστώσεων 130 δισεκατομμύρια στις τοπικές τράπεζες που θα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί αυτό το κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εάν αυτό το κεφάλαιο υποστεί κούρεμα, σημαίνει ότι η ίδια η δυνατότητα δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα γίνει πιο ακριβή. Δηλαδή θα αναγκαστούμε για λόγους ε, ε ρυθμιστικούς, για τήρηση του ρυθμιστικού πλαισίου, να αυξήσουμε το δικό μας κεφάλαιο ε, ε για λόγους φερεγγιότητας, τη δικιά μας πιστοτική επάρκεια. Που σημαίνει ήδη φέτος και θα είναι η πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια που θα έχουμε κάποιες επιτυχίες, δηλαδή που για πρώτη φορά θα αυξηθεί η απασχόληση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, κατά πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια ε, δεν θα αυξηθεί η ανεργία, θα μειωθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τουλάχιστον κινούμαστε προς μια σωστή κατεύθυνση. Τώρα, έρχομαι στο ερώτημα του κύριου Κάλβιν. εάν χρειάζεται μια ειδική εκθέση από το ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε την δανειοδότηση δραστηριοτήτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω θα ήταν σκόπιμο να το να ταιριάξει, να έρθει την ίδια στιγμή με την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση. Λίγους μήνες πριν, ε, για πρώτη φορά, παρουσιάσαμε μια έκθεση δραστηριοτήτων που δείχνει ποιε είναι οι δραστηριότητέ μας εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ποιον τρόπο συνδυάζουμε την ε, δανειοδότηση ε, από την τράπεζα μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση κινδύνου της ίδια τη τράπεζα Επενδύσεων. Θέλω να γνωρίζετε ότι για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το να έχει στάτους 3α δεν είναι φετίχ είναι απαραίτητο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να δανειζόμαστε με πολύ χαμηλό κόστος. Και έτσι μόνο μπορούμε αυτό το πλεονέκτημα να το μετακυλίουμε σε εκείνους που συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Είτε αυτές είναι τοπικές αρχές είτε εθνικές κυβερνήσεις. Είναι λοιπόν εργαλείο το, το, το στάτους των 3α. Έτσι το αντιμετωπίζουμε και γι' αυτό το θεωρούμε τεράστια σημασία. Χρειαζόμαστε να έχουμε αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες δανεισμού. Ο κ. Κάλβιν αναφέρθηκε στο ζήτημα του blending, δηλαδή την χρήση έξυπνων συνδυασμών επιχορηγήσεων και δανείων προκειμένου να ενδυναμωθεί η οικονομία. Εξετάζουμε τη χρήση νέων εργαλείων, νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για να φτιάξουμε τέτοιου είδους συνδυασμούς. Γιατί με τέτοιους συνδυασμούς μπορούμε να βοηθήσουμε την οικοδομία με πολύ καλύτερο τρόπο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που ε, κατά τα άλλα όλοι ακολουθούν πολιτικές λιτότητας. Ε, επίσης αναφερθήκατε στο σύστημα της καινοτομίας, εξαιρετικά σημαντικό και αυτό. Βασική φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο που η Ευρώπη στο μέλλον να είναι ανταγωνιστική. Αυτό αμέσως αμέσως οδηγεί στην κοινοτομία, στην καταπολέμηση του αποκλεισμού και στη βιωσιμότητα. καταπολέμηση του αποκλεισμού προφανώς αναφέρεται στο, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την, την ε, κοινωνική κατάσταση. Επομένως συζητούμε στο πλαίσιο του νέου ε, πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου διάφορες ιδέες και με την Επιτροπή. Για παράδειγμα, ε, κάποια μικρά χρηματοδοτικά, δανειοδοτικά μάλλον εργαλεία προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να μειώνεται το ρίσκο που αναλαμβάνει κάθε μία από αυτές. Η επένδυση σε μεγάλα οδικά έργα, για παράδειγμα, είναι σημαντική και αυτό το κάνει επί χρόνια η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων. Αλλά η επένδυση στη, στην καινοτομία, σε νέε τεχνολογίε, σε νέε ιδέε είναι ακριβώ αυτό που θα μα κάνει ανταγωνιστικού στο μέλλον. Το γνωρίζουμε αυτό και ακριβώ εκεί θέλουμε να εστιάσουμε. Κύριε Οντή, εσείς αναφερθήκατε στο κεφάλαιο το καταβληθέν κεφάλαιο. Το εγγεγραμμένο είναι 144 δισεκατομμύρια. Το καταβληθέν είναι 21-22 δισεκατομμύρια, το οποίο σημαίνει ο συνολικός μας ισολογισμός είναι περίπου 50 δις, σημαντικός, 500 δισεκατομμύρια. και έχουμε διαφορετική κατάσταση από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Άλλα κράτη-μέλη έχουν στάτους 3α, αλλά όχι. Αυτό πρέπει να, όλους, όλους τους παράγοντες πρέπει να τους συνυπολογίσουμε σε μια εξίσωση έτσι ώστε να ε, τελικά το αποτέλεσμα να είναι μια ε, φερέγγια τράπεζα. Στο που κάναμε λοιπόν φέτος με την αύξηση κεφαλαίου ήταν σταδιακό από πέρσι και τις αρχές αυτού του έτους και η επέκταση των πιστοτικών μας δραστηριοτήτων ήταν κατά 40%. Εάν μας το επιτρέψουν οι συνθήκες θα το ξανακάνουμε. Συζητάμε τις λεπτομέρειες, αλλά θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η αντικυκλική δανειοδότηση και τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό μας ζητούν τα κράτη-μέλη. Μα ζήτησαν να γίνει αύξηση κεφαλαίου έτσι ώστε εμείς να λειτουργήσουμε αντικυκλικά. Όσον αφορά τώρα τι μακροπρόθεσμε επενδύσεις. Προφανώς συνεισφέραμε και στην κατάρτιση του πράσινη βίβλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Είμαστε ιδιαίτερα ενεργό μέλο αυτή τη σε αυτόν τον τομέα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί. Έτσι μόνο μπορεί να μειωθεί, όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, έτσι μόνο μπορεί να μειωθεί η εξάρτηση από τον τραπεζικό τομέα. Και να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης άλλων πηγών ε, χρηματοδότησης, άλλων επενδύσεων, επενδυτών, ε, ασφαλιστικών ταμείων, που θα επενδύσουν στην πραγματική οικονομία. η τράπεζα λοιπόν ασχολείται με αυτό το θέμα έντονα και προφανώς ε, η Επιτροπή θα προωθήσει την, πρωτοβουλία μέσω της Πράσινης Βίβλου. Ε, έχω ένα ακόμα σημείο να αναφέρω, αν ξέχασα κάτι θα μου το θυμίσετε, το ζήτημα της εποπτείας. Επί της αρχής δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με οποιαδήποτε μορφή εποπτείας μπορεί να συνειφέρει στους κοινούς μας στόχους. Βέβαια, από τις συνθήκες Ρώμης προβλέπεται ε, η νομική και ρυθμιστική ε, τα νομικά και ρυθμιστικά στοιχεία που διέπουν τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αλλά έχουμε ένα ολόκληρο σύστημα εποπτείας. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία αριθμιστική αρχή που να εποπτεύει την Ευρωπαϊκή, μας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σαν να επρόκειτο για εμπορική ε, τράπεζα. Υπάρχει η ΟΠΑ που μας ε, εποπτεύει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επεκτείνει τις δραστηριότητές της και πρέπει να δούμε εάν αυτό θα έχει επιπτώσεις για δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το δικό μας, αλλά ε, είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε αυτό και το έχουμε πει και στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, Έχουμε την εποπτεία από την ε, Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου. Κάθε μήνα υποβάλλουμε ε, έκθεση ρευστότητα. Έχει δημιουργηθεί μια νέα επιτροπή ελέγχου με σημαντικές αρμοδιότητες. Αυτή δημιουργήθηκε με την ε, συνθήκη της Λισαβόνας που αναφέρεται στις βέλτιστες πρακτικές στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Επίσης το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει τις δραστηριότητες της τράπεζας μας Οποτεδήποτε οι δραστηριότητε μα αυτέ συνδέονται με άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο συμβαίνει πολύ συχνά. Είτε πρόκειται για χρήση άλλων χρηματοδοτικών ε, μέσων, ε, δηλαδή blending, είτε πρόκειται για ε, άμεση δανειοδότηση, τότε πάντα το ελεγκτικό συνέδριο επιβλέπει τη, τη, τη, τη δράση μας. Επίσης, ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής και το Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης, όλα ε, εποπτεύουν την τράση μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι ένα συνδυασμός ε, συστημάτων. Επίσης έχουμε ένα σύστημα υποβολής ε, ε, ενστάσεων. Σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τις διάφορες ενστάσεις. Θα διαπιστώσετε ότι περισσότερες από αυτές ε, επιλήθηκαν φιλικά. Ορισμένε έφτασαν στον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή. Θα έλεγα λοιπόν ότι συνολικά υπάρχουν πολλά ε, κομμάτια στο παζλ της εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή, Τράπεζα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πει εμείς θα θέλαμε να μπορούμε να εποπτεύουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπως και τις ε, τράπεζες των κρατών μελών. Εάν αυτό είναι ο, ο κατεύθυνση προς το οποίο θα κινηθούμε, εμείς είμαστε ανοιχτοί και θα το δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας κάλυψα. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Σιγητή, ο οποίος ήταν σε ψηφοφορίες ε, στην Επιτροπή Μεταφορών να τονίσω πως ε, το συζητήσαμε εδώ αλλά και σε άλλες επιτροπές, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, στην Ολομέλεια. Θέλαμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει περισσότερα πράγματα για τη χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, γιατί ειδικά αυτές είχαν προβλήματα με την πρόσβαση στην χρηματοδότηση ειδικά στις χώρες της κρίσης και μετά βεβαίως η κατάσταση επιδεινωνόταν αυτομάτως. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και ευχαριστώ και τον πρόεδρο τον κύριο Χωά. Ε, μας ε, δεχτήκατε βεβαίως και στο Λουξεμβούργο. Να ρωτήσω ποια άλλη θέλουν τον λόγο εκτός από τον εισηγητή. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Μαρινέσκο όμως. Σας ευχαριστώ. Ε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα, όπως ξέρετε το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή Μεταφορών, όπου είμαι τακτικό μέλος και ψηφίσαμε τα δικαιώματα των αεροπορικών, τα δικαιώματα όλων ημών δηλαδή. Βεβαίως θα έχουμε όλοι δικαιώματα αλλά θα κλείσουν οι εταιρείε αν να πληρώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ακούγοντας τον κύριο Κνάπεν συνειδητοποίησα πως ε, υπόθηκαν σχεδόν τα πάντα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το ε, Είστε μια ευρωπαϊκή τράπεζα, δηλαδή πρέπει να εστιάζετε στην Ευρώπη και ειδικά στις χώρες που έχουν δυσκολίες, γιατί εκεί πέρα χρειάζεστε περισσότερο και είστε επενδυτική τράπεζα, δηλαδή πρέπει να επενδύετε, να δημιουργείτε θέσεις εργασίας και ειδικά ε, στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άρα εκεί πρέπει να δώσετε βάρος. Οπότε, αν όχι τώρα, στο μέλλον μπορείτε να μου στείλετε μία απάντηση σε ένα ερώτημα. Πόσες θέσεις εργασία δημιουργήσατε πέρσι με τις δραστηριότητες σας, ή τα τελευταία τρία χρόνια ας πούμε. Σας ευχαριστώ. Γιάν Μουλτερ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ γιατί έρχονται συχνά εδώ πέρα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, παρά το ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την εγγύηση μόνο 10% του κεφαλαίου σας, μας κακομαθαίνετε λοιπόν. Δύο παρατηρήσεις έχω. Και ο κ. Κνάπεν το είπε. η ελκυστικότητα της τράπεζας σας είναι τα χαμηλά επιτόκια και μπορεί να τα προσφέρει γιατί έχει το 3α και την εγγύηση των κρατών μελών. Αλλά το ένα κράτος μέλος μετά το άλλο χάνει την αξιολόγηση 3α και ανησυχώ για το πώς θα επηρεαστεί η τράπεζα. Ακόμα και στην Ολλανδία χάσαμε. Νομίζω πέσαμε κατά ένα βαθμό πριν από 10 μέρες. Δεν θέλω να σας αφορά τις εξωτερικές ε, επιχειρήσεις. Κάποια πράγματα κάνετε μέσω του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου, αλλά συνεργάζεστε και με άλλες τράπεζες. Την Παγκόσμια Τράπεζα, την Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων, την Αφρικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα κτλ. Αυτές έχουν διαφορετικά συστήματα ελέγχου και μια που ανησυχούμε εμείς για τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, το σύστημα αυτό πώς συνεργάζεται με τις άλλες ε, τράπεζες. Θεωρείτε πως ε, τα συστήματα των τραπεζών αυτομάτως είναι τέλεια ή υπάρχουν άλλοι ελεγκτές εκεί. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε με τον προπολογισμό. Όταν δίνουμε κάτι στον ΟΗΕ ή στους οργανισμούς του ΟΗΕ είναι δύσκολο να δούμε πού πάνε τα λεφτά. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλο συνάδελφος θέλει το λόγο. Όχι. Έχετε το λόγο λοιπόν. Ναι, σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Μαρινέσκο, για την παρέμβασή του. Βεβαίως και θα επανέλθω όταν αναφέρομαι σε τέτοια στοιχεία προτιμώ να προετοιμάσω προσεκτικά την απάντησή μου. Θα σας απαντήσω όμως στην ερώτηση που κάνετε. Κάναμε πολλά πάντως τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε κάνει πράγματα, αλλά δεν θέλω τώρα να απαντήσω περίπου, ούτε να μαντέψω την απάντηση. Θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα αφού προηγουμένως εξετάσω τα στοιχεία. Κάτι άλλο. Όταν οι μέτοχοι είναι αυτοί που τελικά εγγυώνται την τράπεζα, το κεφάλαιο της τράπεζας και βεβαίως αυτοί χάνουν το τα 3α βεβαίως υπάρχει επίπτωση και στην τράπεζα αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά τη δυνατότητα μόχλευσης. Βεβαίως αν όλες οι χώρες έχουν 3α, είναι πολύ ε, μεγαλύτερες οι δυνατότητες χρηματοδότησης, γιατί είναι μεγαλύτερες οι δυνατότητες μόχλευσης. Όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να υπάρχει πολύ σωστή ε, διαχείριση κινδύνου. Και νομίζω ότι η τράπεζά μας έχει καλή πολύ καλή θα έλεγα φήμη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Αν κοιτάξετε τις επιδόσεις μας, Είμαστε εξαιρετικά επιτυχημένοι γιατί είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και συντηρητικοί στην προσέγγιση μας. Τι ακριβώς κάνουμε λοιπόν, βεβαίως και συνεργαζόμαστε και με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κάνουμε συμβάσεις συνεργασίας και βεβαίως ε, πολύ συγκεκριμένα κατανέμουμε τους τομείς ε, αρμοδιότητας των ΜΕΝ και των ΔΕ. Είμαστε μια τράπεζα επενδύσεων και φυσικά πολλές φορές συνεργαζόμαστε με την Παγκόσμια Τράπεζα όταν πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς, για κυβερνήσεις και υπογράφουμε συμβάσεις μαζί τους. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό τμήμα και εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αναπτυξιακές τράπεζες κτλ όλο και περισσότερο προσπαθούμε να συνδυάσουμε τον τρόπο εργασία μας και τα συστήματα. Και μια μεγάλη καινοτομία είναι το θέμα της πρωτοβουλίας ε, για την διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια και τη διαφάνεια. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια και αν κάποιος γνωρίζει τα σωστά συστήματα και εμείς είμαστε σε θέση σήμερα να τα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφάνεια. Υπάρχουν σήμερα μηχανισμοί και συστήματα τα οποία χρησιμοποιούμε για όλους αυτούς που θέλουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματά μας και να τα μετρήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κνάπεν για τις απαντήσεις που δώσατε. Βλέπω ικανοποιημένο και τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε για τις απαντήσεις λοιπόν που μας δώσατε και προσβλέπουμε στην επόμενη συνάντηση που θα έχουμε μαζί σας εδώ στην Επιτροπή Ελέγχου του Προβλήσμου. Νομίζω ότι ελακληρώσαμε και με αυτό το σημείο. Σας εύχομαι και εσάς. Καλά Χριστούγεννα και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αφορά το θέμα της στήριξης της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Βλέπω ότι είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι της Επιτροπής. Καταρχήν όμως θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βέσπερκ από το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω αυτή την ειδική έκθεση του Ελληνικού συνεδρίου για την στήριξη σε ένα ευάλωτο όπως λέμε κράτος, τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Τι ακριβώς εννοούμε. Εννοούμε ε, κράτη στα οποία μία από τις βασικές θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η σωστή η χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να ε, καθοδηγεί την αναπτυξιακή βοήθεια. 500 εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν σε περιοχές ε, που γνωρίζουν έντονες συγκρούσεις και βία και παρόλα τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας η χρηματοδότηση, η αναπτυξιακή βοήθεια παραμένει πολύ χαμηλή. Και βεβαίως βρίσκονται πολύ μακριά χώρες αυτές από την υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας. Σήμερα βλέπουμε ότι χρειάζεται πολύ σοβαρή βελτίωση η διακυβέρνηση στις χώρες αυτές. Ο έλεγχος που έγινε όσον αφορά την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό εξέτασε τις ανάγκες καθώς και την υλοποίηση των στόχων όπως έχουν σχεδιαστεί. 60 προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας, της μεταρρύθμισης της, των δυνάμεων ασφάλειας, ηλεκτρονικά συστήματα. Από το 2003 το 2011 η συνολική αξία αυτών των προγραμμάτων ήταν 400 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι εδώ ουσιαστικό να υπογραμμίσουμε ότι βεβαίως ε, ο έλεγχος έγινε σε παλαιότερα και νεότερα προγράμματα, έτσι ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα αυτών. Διαλέξαμε τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, καθότι αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για μία από τις πιο ευάλωτες χώρες, πιο ασταθείς χώρες, και έναν από τους εταίρους αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2003 στο 2011 το ποσό της αναπτυξής βοήθειας φτάνει τα 9 δις. Και διαπιστώσαμε ότι ενώ υπήρχε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναπτυξιακής βοήθειας στο τομέα το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό για την κάλυψη αναγκών σε όλους αυτούς τους τομείς και την το... κάλυψη των αδυναμιών, μόνο το 50% των ε, προγραμμάτων θα φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα με αργούς ρυθμούς ανάπτυξης των προγραμμάτων και η βιωσιμότητα είναι ένας στόχος που πολλές φορές δεν φαίνεται να είναι ρεαλιστικός. Κάποιες από τις δυναμίες μπορούν να εξηγηθούν από κάποια πολιτικά στοιχεία. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχει ένας σχεδιασμός ασαφής, μη φιλόδοξος, που μπορεί να εξηγήσει επίσης τα πολύ έλλειπη αποτελέσματα, έλλειψη πληροφοριών και επαφών. Η Επιτροπή επίσης δεν χρησιμοποίησε όλες τις δυνατότητες για την δέσμευση των εθνικών αρχών έτσι ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση των δράσεων. Οι συστάσεις μας λοιπόν είναι οι εξής. Πάντα σε σχέση με το πρόγραμμα δράσης για την αναπτυξιακή βοήθεια, να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των κοινοτικών κονδυλίων. Πρώτον, η Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει τη στρατηγική συνεργασίας, καλύτερη γεωγραφική κατανομή στις επαρχίες και με το να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ε, απολογισμό από μέρους των εθνικών και κυβερνητικών αρχών. Δεύτερον, καλύτερη δέσμευση και αξιολόγηση κινδύνου από μέρους της Επιτροπής έτσι ώστε να είναι πιο ρεαλιστική η στόχη των προγραμμάτων για να υπάρξει μεγαλύτερη απορρόφηση πόρων. Καθότι βλέπουμε ότι υπάρχουν αδυναμίες στην εθνική διοίκηση, διαφθορά, χρειάζονται καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να έχει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των στόχων όπως έχουν σχεδιαστεί και της ε, πραγματικότητας, του τι δηλαδή μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη. Επίσης, χρειάζονται περισσότερη δέσμευση των εθνικών αρχών έτσι ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα. Υπάρχουν οι εταίροι των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, των κοινοτικών υπηρεσιών που θα πρέπει να δεσμευθούν όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων, τις προϋποθέσεις και θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση της συμμόρφωσης αυτών των εθνικών ε, αρχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει επίσης να μπορεί να ανταποκριθεί με έναν τρόπο έγκαιρο και βασιζόμενη βεβαίως στην αρχή της αναλογικότητας. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι απαιτητική, να δείξει κατανόηση και να μπορεί να επέμβει εκεί που αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατευθύνουμε τις ε, τοπικές αρχές σε μια καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου των αποτελεσμάτων, κάτι που σαφώς θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας και βεβαίως θα πρέπει να οδηγήσουμε σε περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σωστή στιγμή, καθότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επαναξιολογήσει για την περίοδο 2014-2020 αυτά τα προγράμματα. Οι συστάσεις μας λοιπόν θεωρώ ότι ε, είναι εξαιρετικά επίκαιρες έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογηθεί σωστά η ανάγκη για την μελλοντική χρηματοδότηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέσπερκ. Ο εισηγητής Μπάρτ Στάις έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα να ευχαριστήσω το αρμόδιο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά οπωσδήποτε και τους συνεργάτες του, τους ελεγκτές ε, που έγραψαν αυτή τη σημαντική ειδική έκθεση και πραγματικά έχουμε πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και δεν πρέπει βεβαίως ε, να το θεωρήσουμε κάτι το δευτερεύον πως η δουλειά που γίνεται στο Κονγκό γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ τα τελευταία τρία χρόνια έχω πάει δύο φορές στο Κονγκό. Ως Βέλγος βεβαίως ε, αντιλαμβάνεστε πως ε, ε, υπάρχουν και άλλοι δεσμοί οικογενειακοί και ιστορικοί και Βεβαίω ήμουν ε, και στις ε, προεδρικές εκλογές, μία εβδομάδα στο Κίβο και στο Μπουκάβο. Είδα το τι συνέβη εκεί πέρα, πόσο δύσκολη, όπως είπα, είναι η δουλειά που γίνεται και είχα επαφές ε, με την Επιτροπή εκεί πέρα και τον τότε πρέσβη, τον κύριο Ρίτσαρτ Ζίνγκ, ο οποίος μας εκπροσωπούσε Πρέπει λοιπόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι συνθήκες. Είναι πολύ δύσκολη, όπως είπα, η δουλειά. Αλλά, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, θεωρώ πως η υπηρεσία εξωτερικής δράσης ε, και η Κομισιόν θα μπορούσαν να έχουν δώσει πιο συγκεκριμένες απαντήσεις Εν τω μεταξύ μέσω του Χένκ Πρίμελ ήρθα σε επαφή με τα άτομα της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής ε, Δράσης και μου είπαν κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα να συμπεριλάβω στην έκθεση αλλά βεβαίως θα μπορούσαν όπως είπα να είναι πιο συγκεκριμένοι σημεία τριβής είναι όπως είπα η ερεσιμότητα και ο διάλογος ε, και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα έπρεπε ίσως να προσπαθήσουμε να δώσουμε περισσότερη βοήθεια επιτόπου μέσω των ΜΚΟ. Εγώ διαπίστωσα πως εκεί πέρα όπου δραστηριοποιούνται ΜΚΟ, κογκολέζικοι ΜΚΟ που συνεργάζονται με άλλες ε, με άλλους ΜΚΟ από την Ευρώπη, το αποτέλεσμα συχνά είναι καλύτερο ή πιο προσανατολισμένο θα έλεγα καλύτερα στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Κατόπιν βλέπουμε πως ε, μιλάμε για μεγάλα έργα σε μεγάλο βαθμό ε, τα οποία χρηματοδοτούνται από πολλούς ε, δωρητές. Θεωρώ πως όταν στο μέλλον προκύπτουν τέτοια μεγάλα έργα, ο έλεγχος, ο συντονισμός ε, θα έπρεπε να είναι κάπως πιο κεντρικός από την Κινσάσα σε συνεργασία με την κυβέρνηση βεβαίως γιατί πρέπει και αυτοί να το νιώθουν δικό τους έτσι όταν κάνουμε κάτι και μιλάμε για αναπτυξιακή συνεργασία αλλά μπορεί νομίζω όπως είπα να δοθεί ένας ρόλος στην Κινσάσα στους ανθρώπους της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης εκεί πέρα σε συνεργασία με την κυβέρνηση ε, νομίζω κάτι θα έχει κάποια θετικά αποτελέσματα πέμπτον πρέπει να υπάρξει υπερτέρω διάλογος με τους διεθνείς εταίρους μας που είναι παρόντες στην χώρα η Κίνα έχει μεγάλη παρουσία, δεν μπορεί να διασχίσει κανείς τη χώρα χωρίς να δει εργοτάξια όπου δουλεύουν Κινέζοι. Κινέζικες εταιρείες με Κινέζους εργάτες και πονάει κανείς να βλέπει να φέρουν εργάτες από την Κίνα. Χάνονται ευκαιρίες. Αλλά πρέπει να έχουμε κάποιον διάλογο με τους Κινέζους, με τους λοιπούς εταίρους μας ε, της διεθνούς συνεργασίας και να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος των όσων συμβαίνουν στην πλευρά της διοίκησης. Έκτον, η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει, το κάνουν ήδη, αλλά πρέπει ακόμη περισσότερο να παίξουν έναν ρόλο προληπτικού διαλόγου με τις αρχές της λαϊκής δημοκρατίας να χρησιμοποιήσουν ό, όλους τους ε, διπλωματικούς διάβλους για να υπάρξει πραγματικός σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών. Το επόμενο είναι δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι, η αιρεσιμότητα. Πώς ως ένας σημαντικός δωρητής φροντίζεται αυτά τα οποία δίνεται ε, να χρησιμοποιούνται όπως πρέπει. Στον διάλογο που είχαμε την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ακούσα και βεβαίω προκύπτει αυτό και από τις συμφωνίες που έχουμε με τις χώρες ΑΚΕ, από τις συμφωνίες Κοτονού, πως ε, υπάρχει μια ολόκληρη φιλοσοφία και η Κομισιόν και η Υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης ε, ε, ακολουθούν μια πολιτική σταμάτα ξεκίνα ανάλογα με την πρόοδο που υπάρχει. Πρέπει, λέει η Συμφωνία του Κοτονού, να γίνει περισσότερη δουλειά μέσω πολιτικών συμφωνιών, μέσω εταιρικών σχέσεων. Οπότε θα μπορούσε εδώ πέρα η Κομισιόν να σκεφτεί ποια μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε ακριβώς ε, η πολιτική αυτή στόχοι να μην εμποδίζονται από την αιρεσιμότητα, πώς να το πω, τις προϋποθέσεις. Θα μπορούσαν εδώ πέρα λοιπόν να έχουν κάποια, κάνουν κάποια πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορεί να μπουν μετά στις συστάσεις του ψηφίσματος. Αυτές ήταν οι προσωπικές μου παρατηρήσεις. Έχω υποβάλει το σχετικό έγγραφο εργασίας. Υπάρχουν πέντε σημεία που είναι συστάσεις που θα μπορούσαν να μπουν στην έκθεση της απαλλαγής και στις ειδικέ εκθέσεις. Αντιλαμβάνομαι από την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πως συμφωνούν με τις περισσότερες από αυτές τις συστάσεις. Θα ήθελα να πω επίσης τους συναδέλφους Ε, κάποια πράγματα στα οποία θα ήθελαν μια κάπως διαφορετική απόχρωση η Κομισιόν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εκεί πέρα που λέω παραδείγματος χάρη στο σημείο 1α για όλες τις περιφέρειες και τα λοιπά. Ε, αναφερόμαστε βεβαίως στον Ανατολικό Κονγκό που υπάρχουν οι συγκρούσεις ε, οι οποίες τώρα είναι σε κάποια ύφεση αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα ήθελα εδώ πέρα κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες, ε, κάποια, κάποιες περισσότερες λεπτότερες αποχρώσεις αν θέλετε. Επίσης για το περιβάλλον, ε, την βιώσιμη ανάπτυξη και στο σημείο 4α όπου χρησιμοποιώ τον ε, όρο όρη προϋποθέσεις Ε, μπορεί να αντικατασταθεί νομίζω από την έννοια των στόχων έτσι ώστε η διατύπωσή μας να ευθυγραμμιστεί με αυτά τα οποία λένε οι συμφωνίες Κοτονού. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ακούσω τώρα τους συναδέλφους και τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ, κύριε Στάς. Η κυρία Βάιλερ έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Βέστερ και τον εισηγητή. Θα ήθελα να βασιστώ και στις δύο αυτές παρουσιάσεις. Καταρχήν, η ειδική έκθεση του Ελεκτικού συνεδρίου είναι πάρα πάρα πολύ επικριτική, αλλά προφανώς είναι και σωστό. Βασίζομαι μόνο σε αναλύσεις, σε στοιχεία, σε εκθέσεις που διαθέτουμε, αλλά πιστεύω ότι είναι σωστές αυτές οι επικρίσεις. Ο κύριος Βέσμπερκ έχει εκφράσει εδώ μπροστά μας και κάποιες πολύ αυστηρές παρατηρήσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, λέγοντας ότι τα προγράμματα στο Κονγκό δυστυχώς δεν είναι βιώσιμα. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση ότι οι ιδέες και οι προτάσεις που εμπνέουν μια τέτοια αναπτυξιακή πολιτική, πολιτική αναπτυξής βοήθειας, θα πρέπει να διακατέχονται από βιωσιμότητα. Επίσης πιστεύω ότι αυτό που ονομάζετε εσείς εσωτερική εθνική δέσμευση Βεβαίως και θα πρέπει να ενισχυθεί. Είναι μια προϋπόθεση και ξέρουμε ότι άλλες εμπειρίες μας δείχνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Βεβαίως χρειάζεται και μεταρρύθμιση επιτόπου. Αυτό σίγουρα μπορεί να οδηγήσει σε βιωσιμότητα. Καλύτερη συνεργασία. Τι να σας πω. Και εδώ αυτό με ξάφνιασε λίγο. Έχουμε πολλά χρόνια εμπειρίας των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών, αλλά και στα πλαίσια των ε, Ηνωμένων Εθνών το διαπιστώνουμε αυτό. Οι διεθνείς οργανισμοί όντως θα μπορούσαν να συνεργαστούν πολύ καλύτερα από ό,τι το κάνουν. Υπάρχει έλλειμμα, ε, το ξέρουμε σε πολλά επίπεδα καλής συνεργασίας. Και παραδείγματο χάρη αυτό που συμβαίνει με τους Κινέζους, ίσως θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε κι εμείς από αυτό που γίνεται εκεί. Έχω και κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την παρουσίαση του εισηγητή. Δεν τα διάβασα όλα βέβαια, αλλά όσον αφορά την ειδική σημασία που μπορεί να έχουν οι γυναίκες επιτόπου, ιδιαίτερα η αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική αλλά και στην Ασία, οι εμπειρίες που έχουμε μέχρι τώρα μας δείχνουν ότι η στήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, ατομικών επιχειρήσεων που απευθύνονται σε γυναίκες είναι ένας παράγοντας επιτυχίας. Τίποτα τέτοιο δεν είδα στην ε, έκθεση ούτε του ελεκτικού συνεδρίου ούτε του εισηγητή. Επίσης δεν είδα πουθενά, Μπάρτ, να αναφέρει στο θέμα της αποκέντρωσης. Πρόκειται για μια μεγάλη χώρα σε έκταση, όχι σε ίσως πληθυσμό, με 8 επαρχίες, περιφέρειες και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα κέντρα. Καλή διακυβέρνηση, ήταν το δεύτερο σημείο που ανέφερες, Μπάρτ. Βέβαια, η καλή διακυβέρνηση είναι το ευκταίο, αλλά τελικά μακάρι να υπήρχε διακυβέρνηση και βλέπουμε για την χρηστή διακυβέρνηση. Καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαι εδώ και δύο χρόνια. Τι να σας πω, ακούγοντας και το ελεγκτικό συνέδριο και τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου διαπιστώνουμε ότι η διαφθορά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους τοπικούς παράγοντες. Οι επιχειρήσεις οι ευρωπαϊκές που δραστηριοποιούνται επί τόπου ε, το κάνουν χρησιμοποιώντας αυτές τις πρακτικές διαφθοράς. Και έχουμε πολλά παραδείγματα δικών μας επιχειρήσεων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ολοκληρώνω. Βεβαίως και θα πρέπει να περιοριστούμε σε ρεαλιστικές προτεραιότητες, το δικό δίκτυο, το δίκτυο της υγείας, Όμως δεν διάβασα πουθενά την ε, εκπαίδευση. Το νερό βεβαίως και τα ποσοστά, τα νούμερα που είδα όσον αφορά την πρόσβαση στο σύστημα το εκπαιδευτικό είναι πάρα πολύ χαμηλά. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και τις γυναίκες και τους νέους να έχουν εύκολη πρόσβαση στην παιδεία. Το σημείο 5 που ανέφερες, Μπάρτ, εκεί που λες ότι η Επιτροπή θα έπρεπε, όχι δεν θα έπρεπε, πρέπει. Αν θέλουμε να διαπιστώσουμε ποια είναι τα προγράμματα που δεν απορρόφησαν, δεν χρησιμοποίησαν τα κονδύλια, εδώ χρειάζεται να υπάρχει και η επεξήγηση το γιατί είτε γιατί δεν ζητήθηκαν, δεν απορροπήθηκαν τα κονδύλια, είτε για άλλους λόγους. Εμείς θέλουμε εδώ να υπάρχουν οι λόγοι. Ευχαριστώ πολύ και κατά τα άλλα βεβαίως θα στηρίξουμε την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιλερ. Η κυρία Γκρέσλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμένα με εξέπληξε η αυστηρή κριτική του ελεγκτικού συνοδρίου στις εκλογές. Εγώ θεώρησα διεξαγωγή των εκλογών μεγάλη επιτυχία και το ότι κέρδισε κάποιος τώρα ο οποίος δεν θα έπρεπε να κερδίσει. Ε, αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να αμφισβητήσουμε το αποτέλεσμα. Μετά κύριε Βέσπερ να σας πω ότι συζητάνε στους διαδρόμους της Κομισιόν. Εκεί πέρα λένε πως είναι βελγική υπόθεση, δηλαδή ο Βέλγος ε, ε, του ελεκτικού συνεδρίου και ο Βέλγος Επίτροπος ε, μονοπολούν το θέμα. Κοιτάξτε, θα αποτελματωθεί η κατάσταση, αλλιώς και η κριτική δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ε, το Κονγκό από μόνο του είναι ε, από άκρη 4.500 χιλιόμετρα, μεγαλύτερο από ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, έτσι. Αν δίνουμε ένα δισεκατομμύριο το χρόνο για μια έκταση όσο ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι περιμένετε με αυτά τα λεφτά. Όχι η σταγόνα στον ωκεανό, ούτε αυτό δεν είναι. Και εσείς ε, κυρία Βάιλερ μιλάτε και για εκπαίδευση και να φτιάξουμε εκπαίδευση. Τι να σας πω. Εγώ προτιμώ κάτι πιο στοχευμένο, ε, γιατί τίποτα άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε, έτσι. Να σας υπενθυμίσω πως έχουμε μεταξύ 70 και 80 ατόμων. Ε, εντάξει, ε, τι να κάνουνε και αυτοί, τι να πρωτοκάνουν. Ε, πατάμε στη γη, να είμαστε ρεαλιστές. Πέρα δηλαδή από κάποια διακοσμητικά πράγματα δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε με τα κονδύλια που έχουμε εκεί πέρα και με τον τρόπο με τον οποίο ε, δηλαδή με τις δυσκολίες με τις οποίες πρέπει να λειτουργήσουμε. Δεν ξέρω, θα ήθελα να μου απαντήσετε κάτι γι' αυτό και για το ενδοβελγικό ζήτημα. Μάλιστα, ε, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω από τα μέλη της Επιτροπής, οπότε κύριε Βέσπερκ, αν μπορείτε να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Υποθέτω σωστά πως για τη σύνταξη της έκθεσης πήγαν κάποιοι επιτόπου και είδαν τα πράγματα η διεισόμαση. Αλλά πήγατε κι εσείς αυτοπροσώπως και πώς λύσατε τα πρακτικά ζητήματα γιατί τα είπε και η κυρία Γκρέσλε δηλαδή το μέγεθος της χώρας οπωσδήποτε καθιστά και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους ε, δύσκολους και δεν ξέρω ίσως όχι και τόσο ουσιαστικούς Α, ίσως έχουμε σχηματίσει και λάθος εντύπωση, δεν ξέρω. Θα μπορούσατε λοιπόν να απαντήσετε σε αυτά. Thank you, Ευχαριστώ. Ξεκινώ από το ερώτημα του τελευταίου, εάν κάναμε επιτοπία επίσκεψη, πράγματι, για τρεις εβδομάδες βρισκόμαστε στο Κονγκό και επισκεφτήκαμε τέσσερις επαρχίες. Προσωπικά δεν πήγα γιατί δεν γνωρίζω γαλλικά και μάλλον θα ήμουν βαρύδι στην αποστολή. γιατί αναγκαστικά θα χρειαζόμασταν διερμηνέα τα συνεχώς και δεν θεωρήσαμε σκόπιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Έγραψα μερικά από τα ερωτήματά σας και θα τα απαντήσω. Πράγματι, ασκήσαμε κριτική στην εκλογική διαδικασία στις εκλογές, αλλά είναι τελείως διαφορετικό οι εκλογές του 2005-2006 και οι εκλογές του 2011. Οι εκλογές του 2005-2006, όσον αφορά αυτές, επισημαίνουμε ότι τα περισσότερα γράμματα τα οποία υποστήριξαν την διαδικασία, τη διενέργεια των εκλογών ήταν επιτυχή, ενώ αυτό δεν συνέβη το 2011. Απ' την άλλη βέβαια θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το γεγονό και μόνο ότι διοργανώθηκαν εκλογές στο Κονγκό ήταν επιτυχία από μόνο του. Ίσως θα μπορούσαμε να ήταν πιο συγκεκριμένοι και να εξηγήσουμε περισσότερο γιατί επιλέξαμε το Κονγκό, γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα έφτρας της χώρας. Δηλαδή μιας χώρας η οποία παρουσιάζει προβλήματα πολύ ε, χαρακτηριστικά και τυπικά άλλων ε, εύθραυστων χωρών. Μπορούμε να πούμε ότι το χρησιμοποίησαμε ως μια πιλωτική μελέτη. Από την έκθεση και από την παρουσίαση που σας έκανα πρέπει να πω ότι τελικά ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με την κατάσταση στο Κονγκό από ότι υπό συνθήκες θα ανέμενε κανείς. Ωστόσο, αυτά τα προβλήματα ε, είναι πολύ παρόμοια και σε υπόλοιπες ε, και σε άλλες ε, εύθραυστες χώρες και θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια βοήθειας προς αυτές τις χώρες. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διδαχθούμε και από το παρελθόν. Γιατί αυτά, αυτές οι χώρες είναι εξορισμού ε, ένα περιβάλλον και εξορισμού περίπλοκες. Τώρα για το ζήτημα της ερεσιμότητας αυτό είναι περίπλοκο και το γνωρίζουμε όλοι. Η απόφαση, η άποψη του ελεκτικού συνεδρίου είναι ότι όταν γίνεται Διάλογο με κυβερνητικές αρχές μιας εύθραυστη χώρας εν προκειμένου το Κονγκό, το πρώτο πρώτο στοιχείο στον ε, διάλογο είναι ότι ταυτόχρονα θα πρέπει να απαιτούμε και ταυτόχρονα να δείχνουμε κατανόηση. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, αλλά πρέπει να υπάρχει ε, ξεκάθαρο το στοιχείο της αιρεσιμότητας στον διάλογο, γιατί χωρίς αυτό δεν πιστεύω ότι είναι εφικτό να ε, υπάρξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αντιλαμβάνομαι την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία του εγχειρήματο, αλλά είναι πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Yeah. Thank you very much. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις επιπλέον πληροφορίες. Η Επιτροπή. I would like to give the floor to the Commission. Να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Ο κύριος Βερμπέκε. Εγώ είμαι ο διευθυντής και λέγομαι Πιέρα Amiat, υπεύθυνο για την κεντρική και δυτική Αφρική. Διάφορες α, αδύναμες ε, ευάλωτες χώρες υπό την δική μου αρμοδιότητα. Ευχαριστώ πολύ το Ελεγκτικό Συνέδριο για την παρουσίασή τους. Ο Επίτροπος καθώς και η Αντιπρόεδρος Επιτροπής, κυρία Άστον, έχουν πει ότι είναι προτεραιότητα η συνεργασία και η αναπτυξιακή βοήθεια και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε ένα επικοδομητικό διάλογο. Τώρα, όταν μιλάμε για ευάλωτες χώρες, είναι εύκολο να χρησιμοποιήσει κανείς ένα δείγμα όπως το ανέφερε εξάλλου και το ελεκτικό συνέδριο. Δεν είναι εύκολη όμως έννοια για να ορίσουμε και δεν υπάρχει και μια έτοιμη λύση η οποία να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα και να προτείνει και μία μέθοδο αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών των ευάλωτων χωρών. Αυτές οι χώρες έτσι και αλλιώ προτείνουν μια προσέγγιση του ευάλωτου χαρακτήρα. Και η έννοια αυτή για πρώτη φορά έγινε αποδεκτή στο Μπουζάν στην Σύνοδο για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και τη Συνεργασία. Θεωρούμε λοιπόν σήμερα ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε κάποιες διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε στόχους αποδεκτούς από τις δύο πλευρές. Ο εισηγητής προτείνει κάποιους τέτοιους στόχους. Εγώ θα έλεγα προσυμφωνημένους στόχους, δηλαδή πρόκειται για συμβατική, αν θέλετε, προσέγγιση και σχέση μεταξύ των δωρητών και των ευαίσθητων αυτών ε, έδραυτων χωρών. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι συστάσεις του εισηγητή αλλά και του ελεγκτικού συνεδρίου για την καλύτερη κατανομή της στήριξης, της βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να καλύψει όλες τις ανάγκες του Κονγκό, αυτό είναι κατανοητό. Απαντούμε λοιπόν σε αυτήν την επιθυμία λέγοντας ότι χρειάζεται καλό συντονισμός έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη κάλυψη των αναγκών όλης της επικράτειας αυτής της χώρας. Σήμερα μεταξύ των δωρητών υπάρχει συμφωνία για την περίοδο που μας αφορά και φυσικά θα υπάρξει ε, συγκέντρωση της χρηματοδότησης και των προγραμμάτων εκεί που υπάρχουν οι μεγαλύτερες ανάγκες στο Ανατολικό Κονγκό συγκεκριμένα. Τώρα, είμαστε ή δεν είμαστε ρεαλιστικοί όταν θέτουμε τους στόχους και τις φιλοδοξίες. Ναι, μπορούμε να είμαστε ρεαλιστές. Ιδιαίτερα όταν ε, οι στόχοι είναι μετρήσιμοι. Πόσα χιλιόμετρα οδικό δίκτυο, είτε πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν περάσει από τα προγράμματα κατάρτισης ή την ηλεκτροδότηση κάποιων περιοχών. Άλλοι στόχοι είναι πολύ λιγότερο μετρήσιμοι. Παραδείγματο χάρη, πώς μπορούμε να περάσουμε στις χώρες αυτές τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκπαιρέωση δημοκρατικών και δίκαιων εκλογών. Αυτοί οι στόχοι μπορεί να μην φαίνονται φιλόδοξοι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για την αξιολόγηση αυτών των, της υλοποίησης αυτών των στόχων. Παραδείγματος χάρη διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς κτλ. Η συνεργασία με περισσότερους μη κυβερνητικού οργανισμούς, βεβαίως, αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Στην περιοχή όμως, βεβαίως οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να παίξουν ένα πάρα πολύ θετικό ρόλο όσον αφορά την προετοιμασία των ε, εκλογών, θέματα διαφθοράς, καταπολέμησης διαφθοράς, βεβαίως μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Το θέμα όμως είναι πώς μπορούν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. Αν αρκεστούμε μόνο στους μη κυβερνητικού οργανισμούς, καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν θα αναπτυχθεί ένα τοπικό δίκτυο κυβερνητικό, εθνικό, παροχής αυτών των υπηρεσιών, καθότι υπάρχει και το θέμα της βιωσιμότητας και του κόστους αυτών των ε, προσπαθειών. Οι Κινέζοι τώρα. Εγώ έχω επισκεφτεί πολλές φορές την Αφρική. Οι Κινέζοι είναι παντού. Και δεν νομίζω ότι η διακυβέρνηση θα ήταν το πρώτο που θα έβασα στο επίκεντρο της συνεργασίας και του διάλογου μας με τους Κινέζους. Βέλτιστες ε, πρακτικές ε, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επίσης ε, πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφορά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν και το επιλέγουν οι περισσότερες επιχειρήσεις από την Ευρώπη. Αλλά οπωσδήποτε σε κάποιο επίπεδο, στρατηγικό, υψηλό επίπεδο, έχουμε πολύ υποκοδομητικό διάλογο με τους Κινέζους και είναι πιο εύκολο αυτό να γίνει στο Πεκίνο παρά εκεί επιτόπου στην Αφρική. Δεν είναι μόνο όμως οι Κινέζοι δραστήριοι στην Αφρική, υπάρχουν και οι Τούρκοι και οι Μαροκινοί και άλλοι. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θέμα τη σύσταση έτσι όπως έχει προετοιμαστεί. Είναι κάτι που πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να το ξαναδούμε η λέξη «ερεσιμότητα» επίσης το θέμα των κοινά αποδεκτών στόχων στόχων που έχουν συμφωνηθεί από τα δύο μέρη και για τους οποίους υπάρχει κοινή ε, ευθύνη. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, και όσον αφορά την, τις προθεσμίες που θα πρέπει να τηρηθούν για να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία ή για να μην διακοπεί. Ξέρουμε ότι αν ε, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια διατυπώσουμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα δημιουργηθεί μια καλύτερη διαδικασία η οποία θα οδηγήσει σε πολύ πιο απτά αποτελέσματα αυτή η κοινή ευθύνη αν θέλετε που σε πολιτικό διάλογο βεβαίως προϋποθέτει έναν διάλογο με τις χώρες αυτές γιατί χρειάζεται μια πολιτική προσέγγιση όσον αφορά την στοχοθέτηση. Παράδειγμα, οι εκλογές. Δεν θα σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Οι εκλογές, εάν αποφασίσουμε ότι επειδή ο εκλογικός νόμος δεν ε, υιοθετήθηκε, δεν ψηφίστηκε την ημέρα που εμείς είχαμε προβλέψει δεν μπορεί να γίνει δεκτός. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να δεχτούμε τις εκλογές. Δεν θα γίνουν εκλογές, λέει και η Δημοκρατία του Κονγκό. Δεν γίνεται λοιπόν αυτό. Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε άκαμπτοι και γραφειοκρατικοί στην προσέγγιση μας όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν είναι να υπάρχει μια αξιολόγηση αυτής της αρισμότητας η οποία να βασίζεται σε ένα πολιτικό διάλογο στο σωστό επίπεδο εκεί που πρέπει να γίνει το πολιτικός διάλογος. Θέμα της ιδιοκτησίας, όπως είπε η κυρία Βάιλερ, η βιωσιμότητα των ε, προγραμμάτων αυτών είναι κάτι καθοριστικό οι αρχές, η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία βεβαίως, γιατί συνεργαζόμαστε όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων. Ξέρουμε ότι πάνε μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουν ε, εικοσαπλασιάσει τα κονδύλια για τις κοινωνικές δαπάνες. Απ' την άλλη, Βεβαίως βλέπουμε πολύ αρνητικά σημεία όταν βλέπει κανείς τις αμοιβέ κάποιων κυβερνητικών παραγόντων. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να δεσμευθούν οι κρατικές, οι κυβερνητικές αρχές και ο ρόλος των γυναικών. Ναι, αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Μέρι Ρόμπινσον αλλά και τους επιτρόπους. Μέρι Ρόμπινσον που εργάζεται στο... για το θέμα του Κονγκό. Και βεβαίως θέλουμε να στηρίξουμε τις γυναίκες. Υπάρχει και μία πρωτοβουλία για τη βία κατά των γυναικών. Ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει το Κονγκό. 20 εκατομμύρια συν 5 από τη UNICEF χορηγήθηκαν για το θέμα αυτό της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Τώρα τι μπορούμε να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Ναι, πρέπει να δούμε την αποκέντρωση της δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο μη κυβερνητικού οργανισμούς αλλά και τοπική αυτοδιοίκηση αν υπάρχει ή συνδυασμό και των δύο για την απορρόφηση των κονδυλίων. Ολοκληρώνοντας θα σας πω ότι το σχόλιο της κυρίας Γκρέσλε όσον αφορά την συγκέντρωση και τη στοχευμένη βοήθεια. Ναι, βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή μεταξύ των δωρητών σε συνεργασία και με την τοπική κυβέρνηση. Και βεβαίως από του χρόνου οι τομείς στους οποίους θα συγκεντρώσουμε την στήριξή μας είναι η ασφάλεια, μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις αστυνομικές δυνάμεις, τη δικαιοσύνη για να υπάρξει ένα ελάχιστο πλαίσιο προστασία ασφάλεια για τους πολίτες. Δεύτερον, προστασία των φυσικών πόρων, των περιβάλλων και βεβαίως οι υποδομές κατασκευή οδικού δικτύου. Δεν υπάρχει στα διμερή προγράμματα, αλλά σε κάποιες ευάλωτες χώρες, σε χώρες με πολύ μεγάλες αποστάσεις, μεγάλη έκταση, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, που από το ανατολικό σύνορο έως το δυτικό μπορεί κανείς να ταξιδεύει μέρες η ανάπτυξη οδικού δικτύου αποτελεί ε, στρατηγικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε που μακρηγόρησα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ την Κομισιόν. Το λόγο έχει πάλι η συγητής. Η κυρία Γκρέσλε, μήπως θέλει να μιλήσει. Με συγχωρείτε. Αλλά Μόλις έλαβα ένα έγγραφο της κυρίας Μακοβέ η οποία θα ήθελε να το διαβάσει γιατί δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από την χρήση του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου και έχει κάποιες ερωτήσεις. Τι γίνεται με τον συντονισμό μεταξύ κρατών μελών και διεθνούς κοινότητας. Πώς θα γίνει καλύτερη στο 11ο Αναπτυξιακό Ταμείο. Μετά θα ήθελε επίσης να μάθει τι γίνεται με τους μηχανισμούς διαφθοράς που περιγράψατε και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Μετά θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι γίνεται για την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, όπως είπα, από τα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και βεβαίω είπαμε πως ε, υπήρχε μια δέσμευση από τον ε, νυν Υπουργό Δικαιοσύνης να καταπολεμήσει τη διαφθορά και θέλαμε να μάθουμε τι γίνεται πρακτικά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πριν δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της, ε, υπηρεσίας, της εξωτερικής υπηρεσίας, ε, νομίζω ο εισηγητής έχει κάποιες ερωτήσεις. Όχι. Με ερωτήσεις από τους βουλευτές, όχι. Οπότε σας παρακαλώ να τοποθετηθείτε. Είναι ο Διευθυντής Εξωτερικής Υπηρεσίας, ο κύριος Κένφαν Φερβέρκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πρόσωπο την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είμαι επίσης ε, συντονιστής για, για την περιοχή των μεγάλων ε, λιμνών της ε, Αφρικής, οπότε μέρα νύχτα παρακολουθούμε την διαδικασία αυτή περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής. Όπως ε, είπε και η ύπατη εκπρόσωπος και ο Επίτροπος Πίμπαλξ ε, στην επιστολή του στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι και εγώ θα συμφωνήσω με τον ε, συνάδελφο. Απλά θα αναφέρω κάποια ζητήματα χάρη συντομίας. Είναι... Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την έκθεση και νομίζουμε πως είναι αρκετά επίκαιρη γιατί προγραμματίζουμε βεβαίω για το μέλλον αλλά ε, είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή στην περιοχή αυτή της Αφρικής πρέπει λοιπόν να είμαστε συντονισμένοι για να στηρίξουμε αυτές τις εξελίξεις δεύτερον η έκθεση εστιάζεται όπως είπαμε στο ότι ε, η χώρα είναι ευαίσθητη, αλλά βεβαίως ε, πάρα πολύ δύσκολο είναι και το περιβάλλον και βεβαίως ε, βασικό εδώ πέρα είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι, αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Και αυτό δεν πρέπει να μας σταματά από το να Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ε, για να αναπτυχθούν κάποιοι θεσμοί που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες και την ανάπτυξη. Η πρόκληση λοιπόν που αντιμετωπίζουμε ε, όταν εργαζόμαστε στη Σομαλία, στο Νότιο Σουδάν, στην Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία είναι ακριβώς να βρεθεί αυτή η λεπτή ισορροπία. Κατόπιν. Και ο χρόνος έχει σημασία. Οι αλλαγές είναι αργές, ιδιαίτερα στην Αφρική αλλά και αλλού και όταν σημειώνεται κάποια πρόοδος δηλαδή αν καρφόταν σήμερα η έκθεση ήταν κάπως διαφορετική αλλά βεβαίως πρέπει να μαθαίνουμε από τις εμπειρίες μας και οι συζητήσεις που είχαμε σήμερα και τους τελευταίους μήνες νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος για τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Απλά να πω πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει μια τοπική ε, δυνατότητα διοίκησης, κράτους. Δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε αυτό, αλλά μπορούν να βρεθούν άλλοι τρόποι και νομίζω η αποκέντρωση στο Κονγκό είναι βασικό θέμα. Για το ζήτημα του πώς θα υπάρχει αμοιβαία λογοδοσία. Ναι, σας ε, εξήγησαν το πλαίσιο του Μπουζάν. Ε. Δεν έχουμε σύμβαση με το Κονγκό, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας του ΟΗΕ με εθνικές δεσμεύσεις το Κονγκό, αλλά και περιφερειακές. Και γίνεται σημαντική δουλειά στο επίπεδο της Κινσάσα για να ευθυγραμμιστούν αυτά τα οποία κάνουμε ως δωρητές με τις δεσμεύσεις αυτές, έτσι ώστε οι δεσμεύσεις αυτές να μην είναι γενικοί στόχοι, αλλά ξεκάθαροι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που θα πρέπει να επιτύχουν οι αρχές και έτσι θα μπορέσουμε να κινηθούμε από κοινού βήμα-βήμα για να έχουμε σημαντικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, και για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, ε, για τους δικούς τους πόρους Οπότε, έτσι, όχι μόνο η χώρα θα έχει σαφείς στόχους, αλλά και οι δωρητές. Και αν συνεχίσουμε την πορεία αυτή, νομίζω πως έχουμε μια καλύτερη πιθανότητα να, να επιτευχθεί πρόοδος. Βεβαίω δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, η διαδικασία είναι δύσκολη, αλλά αν είμαστε ενωμένοι ως διεθνής κοινότητα, και αν έχουμε όπως είπα επαφές με τις αρχές του Κονγκό είμαστε σίγουροι πως έχουμε αρκετές πιθανότητες για α, να επιτευχθεί η πρόοδος. Όλα αυτά όπως είπαμε κοινή λογοδοσία αυτό το οποίο είπε ο πρόσωπος του εκτικού Συνεδρίου για να είμαστε απαιτητικοί αλλά να δείχνουμε και κατανόηση όλα αυτά ισχύουν πράγματι και θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Ναι, Κοιτάξτε, σαν ειδικό εκπρόσωπος, σαν επικεφαλής αντιπροσωπείας, σαν τι πήρατε το λόγο. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο ειδικό εκπρόσωπος δεν ξέρουμε ακριβώς τι εκπροσωπεί. Με ενδιαφέρει ως τι πήρατε το λόγο. Μπορείτε να απαντήσετε. Δεν είμαι ειδικό ε, εκπρόσωπο. Είμαι διευθυντή της Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Είμαι δημόσιος ε, υπάλληλο, αν θέλετε, ανήκω στην ε, υπηρεσία αυτή, γιατί είμαστε τμήμα της διοίκηση. Αλλά ανήκω στην αποστολή των απεσταλμένων και είμαστε πολύ, αν θέλετε, δεσμευμένοι και έχουμε μια έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτό τους τελευταίους μήνες. Πολύ σύντομα να απαντήσω. που τα έθηκαν μέσω της κυρίας Γκρέσλη όσον αφορά το συντονισμό με τα κράτη όσον αφορά το συντονισμό Υπάρχει ένας πολύ δομημένος συντονισμός επιτόπου στην Κινσάσα και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας όλα αυτά που λέει το ελεκτικό συνέδριο. Ακούμε και τις συστάσεις για να βελτιωθεί ο συντονισμός, αλλά αν θέλετε είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε ήδη. Αυτό που είναι σημαντικό με τον συντονισμό είναι ότι υπάρχουν κάποιες ομάδες τεχνικές εμπειρογνωμόνων που εργάζονται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης και συμμετέχουν στις συζητήσεις και το διάλογο μεταξύ των δωρητών. Καταλαβαίνετε ότι η πολιτική όσον αφορά τους δωρητές μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την προσέγγιση που θα έχουν και σε σχέση με τη συμμετοχή των ε, τοπικών αρχών, της κυβέρνησης επιτόπου. Έχουμε λοιπόν μια πάρα πολύ δραστήρια ομάδα στην ε, Κινσάσα που συμμετέχει, που καθοδηγεί κατά κάποιο τρόπο την δράση τον συντονισμό μεταξύ των δωρητών. Για τη διαφορά, τι κάνουμε και τι θα κάνουμε και στο μέλλον. Βεβαίως, έχουμε το πλαίσιο των Υπουργών Δικαιοσύνης. Δεν έχω δυστυχώς εδώ μαζί μου τις λεπτομέρειες του τι ακριβώς γίνεται επί για την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά αυτό που κάνουμε είναι παρόμοιο αυτό που γίνεται σε άλλες αφρικανικές χώρες, διάλογος με την κυβέρνηση όσον αφορά τις διάφορες ε, διαδικασίες ε, που θα πρέπει να αναλάβει η τοπική δικαιοσύνη, το δικαστικό σύστημα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Αυτό θα συνεχιστεί βεβαίως για την μεταρρύθμιση τώρα στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό είναι κάτι που συνεχίζεται. Και βεβαίως αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορώ να σας απαντήσω πολύ συγκεκριμένα ή στην κυρία Γκρέσλη σε οποιοδήποτε άλλο επιθυμεί. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πάρα πολύ σημαντική και έντονη συζήτηση. Ολοκληρώνει ο εισηγητής. Να είμαι σύντομος. Θεωρώ πως ήταν θετική συζήτηση. Είχαμε μια καλή έρευνα του ελεγκτικού συνεδρίου. Μας έκανε να σκεφτούμε τη συγκεκριμένη περίπτωση μιας έφραυστης ε, χώρας ε, όπως ε, η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκού, να σκεφτούμε ποια είναι τα προβλήματα με τον διάλογο με την ε, Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, αντιληφθήκαμε καλύτερα κάποια πράγματα. Επίσης, καλό θα ήταν νομίζω να ξέρουμε πως η Επιτροπή Αναπτυξιακής ε, Βοήθειας αύριο το μεσημέρι θα συζητήσει αυτό το θέμα την έκθεση του ενεκτικού συνεδρίου ε, που οι συνάδελφοι που ασχολούνται καθημερινά με την αναπτυξιακή βοήθεια θα δουν το τι μπορεί να γίνει στον τομέα αυτών και νομίζω πως ε, και η συνεργασία των επιτροπών μας ε, θα είναι χρήσιμη. Επίσης σημειώνω τις παρατηρήσεις της κυρίας Βάιλερ Επίσης, πράγματι, βεβαίως υπάρχουν ε, αηφόρα έργα. Στο Μπουκάβου ε, υπάρχει ένα έργο γεωργίας όπου είναι πραγματικά υποδειγματικά αυτά τα οποία γίνονται. Δηλαδή η καλλιέργεια δεν είναι απλά η αλλά υπάρχει μία αναδάσωση, φυτεύονται νέα δέντρα για μία αϊφόρο δασοκομεία. Επίσης, οι γυναίκες πράγματι στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες παίζουν κρίσιμο ρόλο. Η παρατήρηση της κυρίας Βάιλερ που λέει καλύτερα να μιλήσουμε για διακυβέρνηση και να αφήσουμε αργότερα την χρηστή διακυβέρνηση. Σωστό, το σημειώνω. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρέσλε για τον Βέλγο Επίτροπο Κοιτάξτε, ήταν και υπουργό εξωτερικών και έχουν μείνει ίσως από τότε κάποια πράγματα Εκρεμή, Αλλά και εγώ νομίζω ήμουν, ήμουν παρόν ε, όταν, ε, ανέλα, όταν έγιναν οι εκλογές ε, και ανέλαβε ο νέος πρόεδρος και η ΕΚΟΒΑΣ βεβαίωσε πως ήταν σωστές εκλογές όχι 100% αλλά σε γενικές γραμμές ήταν ε, σωστή η διεξαγωγή τους. Ε, νομίζω επίσης ε, και στο Κίβου ήταν πάρα πολύ θετικές οι εντυπώσεις. Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, έπρεπε να πάνε πολλές φορές για να καταφέρουν τελικά να ψηφίσουν. Υπήρχαν προβλήματα στα εκλογικά τμήματα, αλλά α, δεν τέθη ζήτημα ανοθείας. Ήταν μάλλον περιορισμένες οι απόπειρες. Οπότε νομίζω πως συνεισφέραμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ λοιπόν την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις παρατηρήσεις τους. Οπότε θα τις λάβω υπόψη και θα προσαρμόσω ανάλογα κάπως τις ε, διατυπώσεις. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ ένα περίπλοκο ζήτημα το οποίο συζητήσαμε σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Βέσπερκ ε, και τους εκπροσώπους της ε, Κομισιόν ε, που απάντησαν με επάρκεια. Ευχαριστώ και τους βουλευτές και έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι στα διάφορα. Πότε φαίνεται. Όχι. Αναβάλλεται για το νέο έτος η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε αυτή ήταν η τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα μέλη της Επιτροπής για την συνεργασία. Ευχαριστώ τους πολιτικούς συμβούλους των ομάδων τους συνεργάτες της ε, Γραμματείας και εννοείται βεβαίως ε, και των υπηρεσιών, την νομική υπηρεσία και οπωσδήποτε στους διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια και φέτος εύχομαι λοιπόν προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, καλά Χριστούγεννα και ευτυχές το 2014. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρίαση.